των κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων. Η οικονομία θα πρέπει να εργάζεται για την κοινωνία, θα πρέπει να συνεισφέρει στην κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τι αξιοπρεπεί θέσει εργασία. Θα πρέπει να αποτελεί το εφαλτήριο από το οποίο τα άτομα και οι οικογένειε μπορούν να σχεδιάσουν με εμπιστοσύνη το μέλλον του. Και ενώ πολλά από τα νομιστικά νούμερα ε, της Κομισιόν είναι ε, σημαντικά. Θέλω να τα αναφέρω. Συνεχίζει να ε, μεγενθύνεται η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και προσφέρει αριθμό ρεκόρ θέσεων εργασίας. Σημειώνουμε πρόοδο για τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, το μερίδιο των ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο αποκλεισμού και ε, έχουν, έχει μειωθεί από το 2017 και υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά είναι θετικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλές σημαντικές προκλήσεις που επιμένουν. Για μένα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι ότι έχουν αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό τα εισοδήματα των νοικοκυριών από το ΕΠ σε μία περίοδο 12 ετών. Αυτό μου δείχνει ότι δεν, ε, είναι, δεν υπηρετούμε πλέον την ένταξη. Αυτό όμως είναι ένα σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και για τους πολίτες. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή και επομένως το μέλλον της η ανεργία των νέων ε, είναι ε, ιδιαίτερα υψηλή, στο 5,6% και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, προσπαθήσει να βοηθήσει, Δυστυχώ υπάρχει υποχρηματοδότηση. Έχουμε μια τεράστια πρόκληση της επισφαλού εργασίας. Δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που θα υποστηρίξω την τροπολογία που καλεί για την απαγόρευση των ε, συμβάσεων απασχόλησης μηδενικών ορών. Επίσης, έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής και το 80% της φροντίδας παρέχεται από άτυπους φροντιστές και το 75% αυτών είναι γυναίκες. Ναι, έχουμε την οδηγία για την εξισορρόπηση ιδιωτική και επαγγελματική ζωή. Ε, Όμω, σε ό,τι αφορά τη γονική άδεια, το μέρο αυτό τη οδηγία είναι αδύναμο και επιτρέπει στα κράτη-μέλη που επιλέγουν ε, να μην κάνουν πραγματική επιλογή για του γονεί. Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα στο ψήφισμα ότι οι κοινωνικέ δεσμεύσει και στόχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου σημαντικοί όσο οι οικονομικοί στόχοι και δεν αποτελούν απλώς τα μέσα για να εγγυηθούμε οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να αποτελούν στόχο αυτό καθ' αυτό. Αυτή η προοπτική υπογραμμίζει την προσέγγιση μας σε όλες τις προτάσεις στην έκθεση αυτή σε σχέση με την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη. Σε αυτή η έκθεση στέλνει ισχυρό μήνυμα στους πολίτες ότι εμείς στο Κοινοβουλίο αναγνωρίζουμε την πραγματική ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μπορούν να κοιτούν το μέλλον με εμπιστοσύνη. Σα. ευχαριστώ όλους που έχετε συνεισφέρει στην έκθεση αυτή. Äh, ευχαριστώ κυρία Σότ, τώρα εξ Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, εξωτνά μέλη, σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σήμερα. Ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό τους καιρούς που ζούμε. Το Συμβούλιο προσδίδει μεγάλη σημασία στο Εξάμεινο και χαίρομαι που ανταλλάσσουμε απόψεις με το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό. Εάν θέλουμε να είναι σημαντική η Ευρώπη στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων, θα πρέπει να παραδώσουμε αποτελέσματα στην ανάπτυξη, στι θέσει απασχόληση, σε ψηλό επίπεδο εκπαίδευση, κοινωνική προστασία και περιβαλλοντική αηφορία. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι είναι θέμα λογοδοσίας για τα κράτη-μέλη. Μέσα από τον εξυγχρονισμό των μεταρρυθμίσεων, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει να βελτιώσει την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συμφωνία για κοινού στόχους είναι σημαντική με άλλα λόγια, η έκθεσή σα δείχνει ότι βλέπουμε αυτό τον κοινό στόχο, αυτούς τους κοινούς στόχους και χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει μαζί σήμερα και, ότι έχετε, ε, και με ό,τι έχετε κάνει πρόσφατα με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ξεκινώντας ε, με ένα θετικό σημείο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία τη Ευρώπη έχει ενισχυθεί, η απασχόληση αυξάνεται, οι επενδύσει ανακάμπτουν και τα δημόσια οικονομικά ε, σημειώνουν βελτίωση. Ωστόσο και σαφώ υπάρχουν και παραμένουν πολλέ προκλήσει. Έχετε εντοπίσει μια σειρά από αυτέ τι προκλήσει στι εκθέσεις σα. Οι μακροχρόνιε προκλήσεις παραμένουν όπως είναι η γύρανση του πληθυσμού, η ψηφιοποίηση και αντικτυπώσει στην απασχόληση, η κλιματική αλλαγή και η μη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων η ανάκαμψη των επενδύσεων παραμένει προτεραιότητα έτσι ώστε να προωθήσουμε μια πιο ρωμαλαία ανάκαμψη και να έχουμε ε, ρυθμό ανάπτυξης μακροχρόνια. Η επέκταση του Ταμείου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις σε ό,τι αφορά την χρηματοοικονομική ικανότητα είναι ένα σημαντικό βήμα προς το να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Ας συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί έτσι ώστε να αυξήσουμε τις ε, κοινωνικές επενδύσεις και το ανθρώπινο κεφάλαιο, να άρουμε ε, τα εμπόδια που παραμένουν και να ε, δημιουργήσουμε ένα πραγματικά ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα. Χρειαζόμαστε τη στήριξη με έξυπνες ευφυείς δημοσιονομικές πολιτικές, δίνοντας σημασία στην μακροχρόνια αδιοφορία του προϋπολογισμού μας. Πρέπει επίσης να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίες έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τις οικονομίες για τα προβλήματα και τι προκλήσεις που μας περιμένουν. Θα πρέπει να παρέχουμε στου νεαρού πολίτες υψηλή ποιότητας εκπαίδευση και να επενδύσουμε στις δεξιότητες που έχουν σήμερα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Καθώς ε, αφήνουμε πίσω μας ε, τις περίοδους κρίσης, ε, το κληροδότημα της κρίσης παραμένει μια σημαντική ανησυχία. Αρκετοί πολίτες είναι παγιδευμένοι σε ένα κύκλο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα να ξεφύγουν. Είναι σημαντικό ζήτημα για την Ρουμανική Προεδρία αυτό. Οι προσπάθειες πολιτικής μας θα πρέπει να προσανατολιστούν προς τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Χρειάζονται, ε, πρέπει να προσανατολιστούν και προς εκείνες τις περιφέρειες και τους τομείς που υφίστανται τις περισσότερες δυσκολίες. Θα πρέπει να ε, σκεφτούμε να βρούμε νέες λύσεις σε νέα προβλήματα, ε, δράτοντας επίσης τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Η συνεργιστική οικονομία είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά δεν μπορούμε να πιστοτρομήσουμε σε τομείς όπως είναι τα δικαιώματα απασχόλησης και τα κοινωνικά δικαιώματα. Οι κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να προσαρμοστούν τις αλλαγές που έρχονται στην αγορά εργασίας και να προασπίσουμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η πολιτική ε, στο περιβάλλον μαζί με το πρασίνισμα της οικονομίας και το πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μπορεί να συμβάλλει πολύ σημαντικά στον ευρύ πολιτικό στόχο της τόνωσης ε, της αηφόρου ανάπτυξης και στη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πλήρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και να παρακολουθούμε προσεκτικά την πρόοδο σε κάθε κράτος μέλος. Θα ε, μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και θα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα βελτιστών πρακτικών για να μάθουμε ένας από τον άλλον. Και μόνο με στενή συνεργασία και σταθερή όθηση ε, των προσπαθειών και τη της ε, ε, ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτά αποτελέσματα για κάθε πολίτη και να ξανακτήσουμε την εμπιστοσύνη σε μια δυνατή ε, και μερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και για τις συνεισφορέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα των εισηγητών σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Για την Κομισιόν τώρα, ο κύριος Δομπρόφσκης έχει πρώτος τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητή Ρωμανική Πρόεδρε, η Ευρώπη θα αναπτυχθεί για 7η συνεχή χρονιά. Η απασχόληση ε, είναι σε ύψη ρεκόρ και η ανεργία σε χαμηλά ρεκόρ και συνεχίζουν να μειώνονται, όπως επίσης και το δημόσιο χρέος. Η στρατηγική μας, με βάση τις τρεις προτεραιότητες μας, επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική υπευθυνότητα, αποδίδει όμως η ανάπτυξη είναι μέτρια και οι κίνδυνοι αυξάνονται. Αντιμετωπίζουμε ζητήματα στο εμπόριο και έχουμε ανησυχίες για την βιωσιμότητα δημοσίων χρεών και τραπεζών σε κάποιες χώρες. Επίσης βλέπουμε σε κάποια κράτη-μέλη να μην συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις. Σε κάποιες χώρες εξακολουθούν να έχουν υψηλή ανεργία, άλλες έχουν έλλειψη δεξιοτήτων και έχουμε διαρθρωτικά ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί και εμποδίζουν την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις. Υπάρχουν επίσης μεγάλες ανισότητες εντό και μεταξύ των κρατών μελών. Οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως η γέννηση του πληθυσμού παραμένουν η γρήγορη τεχνολογική αλλαγή. Αλλάζουν την καθημερινή μας ζωή και την εργασία. Γι' αυτό απαιτείται αποφασιστική δράση. Στο εθνικό επίπεδο χρειάζονται στοχευμένες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη. Πρέπει στους καλούς καιρού να μειώσουμε το υψηλό χρέο και να δημιουργηθούν αποθεματικά. Αυτό δυστυχώ δεν συμβαίνει σε κάποια κράτη-μέλη. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σημειωθεί η πρόοδο στην Τραπεζική Ένωση και τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, αλλά κάποια πράγματα ακόμα πρέπει να γίνουν όπω η μεταρρυθμίση των κεφαλαίων αγορών. Στην συνεδρίαση του Eurogroup την ε, εβδομάδα αυτή συζητήσαμε το πώ θα προωθήσουμε τι μεταρρυθμίσει και τι επενδύσει για να υπάρξει σύγκληση. Η Κομισιόν μπορεί να τροποποιήσει την πρότασή τη ε, προ το σκοπό αυτό. Μόλις δημοσιοποιήσαμε τι αξιολογίε μα για τι οικονομικέ και κοινωνικέ προκλήσει σε όλα τα κράτη-μέλη και τι μακροοικονομικέ ε, ανισορροπίε. Επίση είδαμε του τομεί προτεραιότητα για τι επενδύσει, για να έχουμε καλύτερη λειτουργικότητα των ε, ταμείων συνοχή. Για την Βουλγαρία, Ισπανία, Γερμανία, Κροατία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία βλέπουμε ανισορροπίες ε, στο εμπόριο Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία έχουν υπερβολικές ε, ανισορροπίες. Για την Κροατία πρόκειται για μια βελτίωση, να εξεκολουθεί βεβαίω ε, να έχει κάποιες ανισορροπίες στο εμπορικό ισοζύγιο, αλλά δεν είναι πλέον υπερβολικές και έτσι θα μπορέσει τελικά να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Το ίδιο διαπιστώσαμε και στην Ρουμανία, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πέρσι, οφείλεται σε απώλεια της ανταγωνιστικότητας και διεύρυνση του ελλείμματος ε, τρέχουσων συναλλαγών και κυκλικών πολιτικών. Επίσης επισημάναμε τους προβληματισμούς μας για το ύψος του χρέους της Ιταλίας σε σχέση με το ΑΕΠ ε, και στην Ισπανία πάλι. Αλλά αξιολογήσαμε και τις δεσμεύσεις της Ιταλίας προς την κατεύθυνση αυτή. Γενικά, από το 2011 τα κράτη-μέλη έχουν σημειώσει τουλάχιστον κάποια πρόοδο στα δύο τρίτα των συστάσεων, αλλά όπως είπα επιβραδύνονται οι μεταρρυθμίσεις και για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να απευθυνθούν στην υπηρεσία μας η οποία στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις ε, το έχει κάνει ήδη σε 500 φορές και επιπλέον άλλα εκατοντάδες έργα θα χρηματοδοτηθούν φέτος Καταλήγοντας, αγαπητοί βουλευτές, η προσέγγισή μας μας έχει βοηθήσει να οδηγηθούμε προς την ανάκαμψη και να παραμείνουμε στην πορεία της ε, αηφόρου ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους εισηγητές και να μένω την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τον λόγο τώρα έχει η Επίτροπος κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Υπουργέ, εξότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο συγητές ε, για τις δύο εκθέσεις για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης. Οι θετικές οικονομικές εξελίξεις ε, συνεχίζουν να μεταφράζονται σε δημιουργία θέσεων εργασίας. 240 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μια θέση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός. Ε, η ενεργία είναι στο 6,5% και είναι στο χαμηλότερο μέσα στον αιώνα. Οι άνθρωποι που διατρέχουν κίνδυνο φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώνονται σε ποσοστό και ε, σήμερα είμαστε περίπου στο επίπεδο του 2008. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν ωφελεί όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο. Όπως είπε και η συγγήτρια από την Επιτροπή Επασχόλησης, ε, το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών είναι κάτω από το επίπεδο του 2008 σε κάποιες χώρες και εξακολουθεί να υπάρχει υψηλή ανεργία σε κάποιες περιοχές, υψηλό ποσοστό ανέχειας και σε κάποια κράτη-μέλη υψηλή φτώχεια εντός της εργασίας και ε, αυτά που είπε η κυρία Χάρκη να συνάδουν με τη δική μας ανάλυση. Ε, ε, θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε την ανέχεια εντός της δουλειάς, τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία, ε, στις εργασίες, για τη στέγαση και την ισορροπία μεταξύ ιδιωτική και επαγγελματική ζωή. Το περασμένο φθινόπωρο ε, και στι 27 Φεβρουαρίου δημοσιεύσαμε τι εκθέσει αναχώρα όπου παρουσιάζεται πιο λεπτομερώ η κοινωνική και οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη. Για δεύτερο έτο εξετάζουμε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Οι εκθέσει για τι χώρε μα δίνουν μια ιδέα για το που βρισκόμαστε, για τι προκλήσει ενωπιών μα ε, και αξιολογούν την απάντηση που δίνουν τα κράτη-μέλη σε επίπεδο πολιτικής. Επίσης εξετάζουμε το κοινωνικό scoreboard, τον πίνακα αποτελεσμάτων. Βλέπουμε πρόοδο και στους 14 δείκτε του πίνακα και πρώτη φορά οι εκθέσεις των χωρών αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες επενδύσεων σε κάθε κράτος μέλος και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ο στόχο μα είναι να πετύχουμε μεγαλύτερε συνέργειε και συμπληρωματικότητα μεταξύ των οικονομικών πολιτικών, των μεταρρυθμίσεων και των ε, ταμείων για τη συνοχή και είμαι πεπισμένη ότι με κοινέ προσπάθειε ε, και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και με συμβολή των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα καταστήσουμε πραγματικότητα τον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα για όλου του πολίτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Um- ευχαριστώ. Για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, τον λόγο έχει ο κύριος Κόβατσεφ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ε, η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται στο έκτο έτος ε, ανάπτυξης ως αποτέλεσμα της υπεύθυνη δημοσιονομικής πολιτικής και των επενδύσεων. Το θετικό αυτό οικονομικό περιβάλλον θα πρέπει να μας ενθαρρύνει για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη και όχι να επιβαρύνουμε τις μελλοντικές γενιές με χρέος. Πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν και στις ανάγκες τους. Πρέπει να εστιάσουμε στους παραγόντες κινδύνου που υπάρχουν ακόμα τη γύρα του πληθυσμού και την υπερβολική χρήση των ψυχών πόρων. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θεωρεί ότι απαιτείται μια πιο υπεύθυνη ε, στάση απέναντι στην οικονομία και πιο αποτελεσματική παροχή υγείας ε, που θα μπορούσαν να αποδειχθούν μεγάλη σημασία. Καθώς οι μεταρρυθμίσεις παρακολουθούνται στα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη σκοπιά γιατί ε, τα αποτελέσματα καμιά φορά εμφανίζονται πολλά χρόνια ε, μετά από τις ε, πράξεις σας ευχαριστώ για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης η κυρία Μιχαήλοβα έχει τώρα τον λόγο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Η Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη καλωσορίζει την θετική δυναμική των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, μας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει επίδραση στις θέσεις απασχόλησης και στην αγορά εργασίας. Και συνεπώς πιστεύουμε ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις και από δημόσιες και από ιδιωτικές πηγές. Τα κάτι μερη θα πρέπει να συνεργαστούν για να προσελκύσουν περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, έτσι ώστε να οικοδομήσουν ε, σχέσεις, εταιρικές σχέσεις και να πετύχουν μια συμπληρωματικότητα των μέσων και ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζουμε τις προτάσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα μελλοντικά επενδυτικά ταμεία. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία της στήριξης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα είναι πολύ χρήσιμες για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κυρία Γκαρσία πέρας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Ξέμινο να σταματήσει να είναι εργαλείο που να λέει στις χώρες που πρέπει ε, να δαπανίσουν περισσότερο ή λιγότερο, που πρέπει να εξοικονομήσουν και να πραγματοποιηθεί να ε, υποτελέσει ένα εργαλείο για να εγγυάται την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να να μπορέσουμε να ακούσουμε τι γίνεται πέρα από αυτούς τους τέσσερις τείχους ε, και να κατανοήσουμε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από την πολιτική λιτότητα. Ας ακούσουμε τα εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες που την προηγούμενη Παρασκευή στις 8 Μαρτίου βγήκαν στους δρόμους της Ευρώπης για να ζητήσουν μια πιο δίκαιη, πιο κοινωνική και ισότιμη Ευρώπη. Ας ακούσουμε τους νέους που θα βγουν και πάλι στους δρόμους την επόμενη Παρασκευή και θα ζητήσουν μια Ευρώπη που θα είναι ικανή να δεσμευτεί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πράγματι θέλουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό project, θα πρέπει να περάσουμε από την πολιτική λιτότητα στην πολιτική δίκαιη και ισότιμη ανάπτυξη για όλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ορτασούν, επίση από την Επιτροπή Γυναικών. Πολύ σύντομα. Βρισκόμαστε στις 13 Μαρτίου, πέντε μέρες μετά από τις 8 Μαρτίου, οπότε εκατομμύρια γυναίκες βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν τα δικαιώματά τους και κάνουμε μια συζήτηση για τις ε, προοπτικές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, δυστυχώς δεν άκουσαν να αναφέρονται καθόλου ε, οι επίτροποι, ούτε οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Μόνο μία φορά αναφέρεται αυτή η ε, και εγώ θέλω να παρακαλέσω κάτι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι στην επόμενη θητεία. Κάθε έξι μήνε να έχουμε μία ανάλυση τη οικονομική πολιτική συστάση αναχώρα και μην αναλύουμε ούτε τον αντίκτυπο των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων ε, στα δύο φύλλα. Να μην δούμε πώ μπορούμε να μειώσουμε το χάσμα στι συντάξει ή το μισθολογικό χάσμα. Ε, δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν ελπίζω για την επόμενη θητεία να αλλάξουν ριζικά όλα αυτά τα πράγματα. Äh, äh, Σα ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στου ομιλητές των ομάδων και έχω μία παράκληση. Είναι μακρός και ο κατάλογος ε, των ομιλητών και σας παρακαλώ πραγματικά να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας. Γιατί πέντε ώρα έχουμε τις ε, ψηφοφορίες και γνωρίζετε τι γίνεται από πλευρά θορύβου στην αίθουσα λίγο πριν τι ε, ψηφοφορίε. Δεν είναι και Για το ΕΛΚ τώρα η κυρία Κοσλόφ Καράγεβιτς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροποι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Σκιώδης Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν για την εξαιρετική έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν και για το ύφος των διαπραγματεύσεων που είναι πολύ καλό. Ε, στην έκθεση περιλαμβάνονται νούμερα και δεδομένα, δείχνοντα ότι η κατάσταση τη αγοράς εργασίας ε, σημειώνει πραγματική βελτίωση. Η, μειώνεται η ανεργία, έχουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και όλοι οι οικονομικοί δείκτες είναι στο θετικό. Ωστόσο, όλοι αυτός, αυτός ο πλούτος ε, δεν διανύμεται ισότιμα ανάμεσα σε όλους τους πολίτες μας. Υπάρχει ακόμη ε, ε, μια ομάδα εκατόν εκατομμυρίων φτωχών ανθρώπων. Υπάρχει ένα χάσμα συντάξεων ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες, γύρω στο 40%. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται μια ψηφιακή μεταμόρφωση που θα αλλάξει την ανταγωνιστικότητά μας στον κόσμο. Ωστόσο, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς κλειδιά, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη που ε, δεν έχουν αυτές τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Άρα θα πρέπει να στηρίξουμε ε, μια μελλοντική κινητική ψηφιακή Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, κυρία Αρένα. Ευχαριστώ. Η Δύση Επισκόπηση Ανάπτυξη αποτελεί μέρο του συντονισμού των πολιτικών πολιτικών τη Ένωση στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ξέρετε ότι για του σοσιαλιστέ θεωρούμε ότι αυτό το, το εξάμεινο προσανατολίζεται πάρα πολύ στα οικονομικά ζητήματα και όχι αρκετά στα κοινωνικά. Τι νόημα έχει να δημιουργούμε θέσει εργασία αν είναι κακοπληρωμένε και δεν τι προστατεύουμε. Τι νόημα έχει να έχουμε ισορροπημένο προπολογισμό όταν δεν μπορούμε να έχουμε επενδύσει στην παιδεία, στην κατάρτιση και για την οικολογική μετάβαση. Τι νόημα έχει να έχουμε ανάπτυξη αν ε, αυτή δημιουργεί όλο ένα και μεγαλύτερες ανισότητε στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια ότι οι κοινωνικές και πολιτιστικέ ανισότητε είναι ο κύριος κίνδυνος τη δημοκρατία και εμεί το βιώνουμε σήμερα σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Στην ε, πρόταση που έχουμε σήμερα, βέβαια, οι κοινωνικές ανησυχίες έχουν ε, υποστηριχθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης και θα αναφέρω κάποια παραδείγματα καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση μια σημασία που να δίνεται στι αξιοπρεπεί μισθού. επίσης σημασία στι συλλογικέ διαπραγματεύσει, αλλά και σε μεταρρυθμίσει που να μην είναι ει βάρο τη αλληλεγγύη και τη αναδιανομή του πλούτου. Και θα τελειώσω με τι επενδύσει στην οικολογική μετάβαση και θα επανέλθω σε μια τροπολογία που ήθελε να καταθέσει το ΕΛΚ και θέλει να καταθέσει για ψηφοφορία και αφορά τις συντάξει. Σύμφωνα με το ΕΛΚ η μόνη λύση για να έχουμε αξιοπρεπεί συντάξει είναι να μπορούμε να έχουμε ιδιωτικά συστήματα. Να πω στο ΕΛΚ ότι τα ιδιωτικά στοξιδοτικά συστήματα είναι το κύριο εμπόδιο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες σήμερα δεν υποφελούνται από πυλών ιδιωτικών συντάξεων και να λέμε ότι θα ρυθμίσουμε αυτό το πρόβλημα πρόβλημα με τις ιδιωτικές συντάξεις είναι ότι ενισχύουμε σήμερα την ανισότητα εντός της Ευρώπης απέναντι στις γυναίκες, εις βάρος των γυναικών. Είμαστε λοιπόν κατά αυτές τις τροπολογίες γιατί υπάρχουν και άλλες λύσεις για το θέμα των συντάξεων. Σας ευχαριστώ. Για το ECR ο Πάκετ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Τόμ Φαντεκέντελάρε, τον εισηγητή, για την ενδιαφέρουσα έκθεση. Ε, γνωριζόμαστε εμείς από νέοι ε, ο καθένας πρόεδρος στο κόμμα του και τότε ασχολούμασταν το εάν ε, οι άνθρωποι της γενιάς μας θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Γιατί πολλοί νέοι δεν πιστεύουν πλέον στο κοινωνικό συμβόλαιο όπως το γνωρίζαμε. Οι σημερινές συμβάσεις πληρώνονται από τους εργαζόμενους. Αλλά μέσω της γύρανσης ε, μειώνονται συνεχώς και αυξάνονται συνεχώς οι δαπάνες στο Βέλγιο μιλάμε για μια αύξηση κατά 15 δισεκατομμύρια. Αυτή αφορά αυτή η έκθεση. Ποια μέτρα πρέπει να λάβουμε έτσι ώστε οι νέοι που εργάζονται σήμερα θα ξεζουμιστούν για να μείνουν μετά χωρίς σύνταξη. Απαιτούνται επιγόντως μεταρρυθμίσεις γιατί η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διατηρηθεί και τελικά θα πρέπει ο καθένας να φροντίσει μόνος του για τα γεράματα του. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την άλλη ο κύριος Καλβές Αμπών για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας ακούσετε κυρία Τίσεν. Θα είμαι σύντομος με πολιτικό όρεμα. Λοιπόν, στα ισπανικά. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τελικά σε αυτή τη φοιτεία τονίσαμε το θέμα της ε, κοινωνίας, την κοινωνική έξοδο από την κρίση και κυρίως με το ευρωπαϊκό εξάμεινο που αφορά τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα απασχόληση. Αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα και στην επόμενη θητεία. Δεύτερον, λέμε ότι τα επίπεδα απασχόληση είναι καλύτερα παρά ποτέ. Είναι αλήθεια. Προσοχή όμω να μην ξεχνάμε ότι όταν υπάρχει ε, σημαντικό επίπεδο ανεργία σε ένα κράτο είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η κατανομή τη ανεργία επίση είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και κάτι άλλο, οι ανισότητε ε, Πάρα πολλά πρέπει να κάνουμε για το θέμα των ανισοτήτων. Οι επόμενες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές δεν μπορούν ε, παρά να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση των ανισοτήτων. Και τέλος, δύο πράγματα είναι απαραίτητα για το μέλλον για να πετύχουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Καταρχήν, θα πρέπει να έχουμε μία οικονομική και δημοσιονομική πολιτική συντονισμένη και αυτό θα επιτρέψει την αναδιανομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, θα πρέπει να δεκτούμε ότι χρειάζεται οικονομική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Παραδείγματο χάρη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προσφέρονται επιδόματα ανεργία. Σα ευχαριστώ. Για τους ε, πράσινους, ε, η κυρία Όχι, ένα λεπτό, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτριά μας ε, την Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, βλέπουμε τώρα ότι αποδίδεται μεγάλη σημασία στην κλιματική αλλαγή. Η έκθεση υπενθυμίζει την ανάγκη εξυγχρονισμού απομάκρυνσης από τον άνθρακα των μεταφορών, ε, της ενέργειας και ακούσαμε από το Συμβούλιο ότι έχει σημασία η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Γιατί αν δεν αντιδράσουμε, η οικονομία μας και η κοινωνία μας θα πληρώσουν ένα τεράστιο τίμημα. Καθώς θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Αν σκεφτείτε το κόστος πέρσι πλημμυρών, πυρκαγιών κτλ. Και, και το πόσο κόστησαν στον προπολογισμό, η ανάγκη επένδυσης σε σωστές υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό χρειαζόμαστε δημοσιονομικό περιθώριο για να κάνουμε πραγματικές επενδύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ΓΚΟΕ η κυρία Λόπες Μπερμέχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε άλλη μία ευκαιρία, αλλά οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν να συνεχίσουν να ακούνε τα ίδια. Η λιτότητα ήταν ένα λάθος και μια αποτυχία. Οι πολιτικές διαχείρισης της οικονομικής κρίσης μας οδήγησαν στη μεγαλύτερη αύξηση των ανισοτήτων στην Ευρώπη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το ευρώ έχει μετατραπεί σε μια μηχανή που δημιουργεί κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στις χώρες μας. Και ως αποτέλεσμα αυτής της ε, καταιγίδα ε, αυξήθηκε πάρα πολύ ο θυμός ενός μέρους των πολιτών και υπάρχει μια δυσφορία που απειλεί όχι μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και την ίδια τη δημοκρατία. Και Μπροστά στο προφανέ τη κατάσταση αυτή. οι δικές μα εκθέσει συνεχίζουν να λένε σε εκατομμύρια ανθρώπου που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχεια και αποκλεισμού και φόβου ότι όλα πάνε καλά. Αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν είναι λογικό και φαίνεται πως είναι προφανές, προφανής η έλλειψη ε, ενδιαφέροντος να συνεχίζουν να πιστεύουν ε, σε κάτι τέτοιο. Κάποιες ε, ειδήσει ε, μας δείχνουν αυτό που έχουν καταλάβει οι άνθρωποι ότι δεν συμπεριφερόμαστε σε όλους ε, το ίδιο. Ε, δυστυχώς ε, φαίνεται να εξυπηρετούνται μόνο οικονομικέ οικονομικές ελίτ και πολυεθνικές. Αυτό δεν είναι η ορθή οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. E Από τους ΕΝΕΦ, e ο κύριος Ζέγλιστρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε κάθε θέμα και πρόβλημα πολιτικής, και έχουμε πολλά από αυτά, υπάρχει μόνο ε, μία κατευθυντήρια γραμμή, απόλυτη εξουσία στις Βρυξέλλες και αυτή η εικόνα καθίσταται σαφής και επιβεβαιώνεται εκ νέου με αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο για την οικονομική πολιτική και τον συντονισμό. Στο σχέδιο έκθεσης βλέπουμε ότι το ευρώ οδήγησε σε χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και υψηλότερη ανεργία σε σχέση με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Επομένω, η Ευρωζώνη δεν τα πάει τόσο καλά όσο τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η λύση είναι πολύ απλή. Να αποχαιρετήσουμε το ευρώ και όλο το σύστημα της ε, κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Και τώρα βλέπουμε άλλοι μάλλον θεωρούν ότι ε, η λύση είναι περισσότερη ε, κεντρική διακυβέρνηση. Βέβαια έτσι ε, παρεμποδίζουμε και την ανάπτυξη αλλά και άλλους κοινούς στόχους όπως η βιωσιμότητα, η συμπερίληψη. Όλα αυτά αρκεί να μην υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη. Ευχαριστώ. Als Fraktionsloser, Herr eine Minute. Ο κύριος Παλσό, μη εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Ένας, ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης δεν καταλαβαίνει τι είναι το Ευρωπαίο εξάμεινο. Θα προσπαθήσω να ορίσω ε, τον όρο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδεικνύει τα βασικά νούμερα για τον προπολογισμό ενό κράτου μέλου. Και κάθε Απρίλιο πρέπει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν ένα πρόγραμμα σταθερότητα. Ε, το Συμβούλιο ζητάει διορθώσεις, ε, εκδίδει δηλαδή συστάσεις αναχώρα και κατόπιν ε, εξετάζεται πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό. Ουσιαστικά καθορίζονται δηλαδή ε, οι βασικές παράμετροι του προϋπολογισμού και ένα Εθνικό Κοινοβούλιο μπορεί να κινηθεί μόνο εντός αυτού του πλαισίου. Είναι θέμα ε, κυριαρχίας, διότι τα κυρίαρχα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν πια να λαμβάνουν αποφάσεις για τον προϋπολογισμό τους. Έτσι, προχωράμε προς ένα υπερκράτος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φτάνουμε τώρα στους λοιπούς ομιλητές. Ο κύριος Φέρμπερ, ένα λεπ... 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Επίτροπε, ε, κυρία ε, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου τα ε, μηνύματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, ήταν μάλλον κάπως ζωφερά. Ε, θα δούμε αποδυνάμωση της οικονομίας και το εύρος της ε, πτώσης αυτής θα εξαρτηθεί από τις πράξεις μας, ε, όπως εξαρτάται και από τις πράξεις των τελευταίων ετών που είχαμε ε, πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Θα εξαρτηθεί όμως και από τις πράξεις μας μέσα στους επόμενους μήνες. Ε, κοιτώ τα στοιχεία και νομίζω ότι ε, πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν προετοιμαστεί αρκετά για έναν ε, αρνητικό κύκλο, κύκλο οικονομίας. Η Γαλλία εδώ και χρόνια βρίσκεται στα όρια διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και τα στοιχεία από την Ιταλία δείχνουν μάλλον μια πλήρη αποτυχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιμείνει ε, στην εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα. Βλέπω συνέχεια το ίδιο μοτίβο. Ε, οι εκθέσεις των χωρών είναι καταστροφικές, ε, οι συστάσεις δεν εφαρμόζονται και αγνοούνται οι δημοσιονομικοί κανόνες σε μια οικονομικά πιο δύσκολη εποχή και με το Brexit που θα, μας, θα στοιχήσει στην οικονομία μας θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν είναι διατεθειμένη ε, να ε, πάρει την κατάσταση στα χέρια της θα πρέπει άλλα θεσμικά όργανα να το κάνουν. Σίλβα Περέρα, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για τους προσανατολισμούς της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής γίνονται σε μια σημαντική στιγμή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας και πολλών κινδύνων και για την οικονομική ανάπτυξη μεταξύ άλλων. Η έκθεση που θα εξετάσουμε σήμερα το απόγευμα είναι διαφορετική από την αρχική εκδοχή. Πολλές από τις προτάσεις που παρουσίασε η ομάδα μου έγιναν δεκτές και γι' αυτό με μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι η τελική εκδοχή της έκθεσης αυτής θα υπερψηφιστεί από τη σοσιαλιστική ομάδα. Ο κύριος, ε, ο συνάδελφος, ο εισηγητής δηλαδή, ε, ο Τόμ, ε, συνεργάστηκε θαυμάσια μαζί μας και μας επέτρεψε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Το βασικό μήνυμα του Κοινοβουλίου είναι η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ένωσης, θα πρέπει να περάσει σε μια νέα φάση για να αντιμετωπίσει τη νέα οικονομική κατάσταση. Χρειαζόμαστε μια συντονισμένη δράση για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού. Χρειαζόμαστε επίσης να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της έλλειψης δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη κάνουν περισσότερα πράγματα για την αύξηση της, ε, οικονομίας με περισσότερες επενδύσεις. Φυσικά θα πρέπει να γίνεται χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, θα πρέπει όμως να γίνονται και επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να καταπολεμήσουμε την ανισότητα με κοινωνική ένταξη, με την ε, ενεργειακή μετάβαση, με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και με την ε, συμπερίληψη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή η νέα θεώρηση των ε, διορθωτικών αλλαγών θα πρέπει να προωθηθεί. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της οικονομικής και δημοσιονομικής στρατηγικής και ακριβώς γι' αυτό θα υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ήμουνα κάπως πιο γενναιόδορη απέναντι στον κύριο Περέιρα, ε, αλλά δεν μπορώ να είμαι ακόμα πιο γενναιόδορη. κύριε Χοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη διέρχεται ε, μία ε, θετική συγκυριακά ε, οικονομική περίοδο, όμως αντιμετωπίζει μια θετικη συγκυριακα οικονομικη περιοδο όμω προκλήσεων και αυτή η θετική συγκυρία δεν θα συνεχιστεί επάπειρον. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προκλήσεις όπως η ψηφιοποίηση. Πρέπει να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις να δώσουμε κίνητρα στην οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να καταπολεμήσουμε την ανική ανεργία, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο, να εξομαλύνουμε τις ε, ανισότητες, να επενδύσουμε στην παιδεία. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα είναι προσαρμοσμένα στην αγορά εργασίας. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, στο πλαίσιο ε, του μηχανισμού μακροπροληπτικής προστασίας που αναφέρεται, θέλουμε και εξετάζουμε την ε, ε, ε, εποπτεία ορισμένων χωρών για το 2019. Η Πολωνία δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία χωρών γιατί είναι ισχυρή σήμερα. Αυξάνεται η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή και είναι και πολύ θετική. Ο κύριος Σαφχάουζερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε βάλει το ένα πόδι σε έναν καταψύκτη στους μείον 250 βαθμούς και το άλλο σε έναν φούρνο 100 ε, στους 100, μπορεί τέλο πάντων να είναι ε, θετική, τέλο πάντων καλή η θερμοκρασία εν γέννη, γιατί βρίσκεστε και πάλι στους 27 βαθμούς ε, Κελσίου, α, τελικά όμως θα πεθάνετε. Αυτό συμβαίνει και με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Βλέπουμε ότι ακόμα δεν, έχει καταφέρει να, δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στα επίπεδα ανάπτυξη που είχαν παλαιότερα. Η Γαλλία το κατάφερε, αλλά χάρη σε ε, ελλείμματα που πλέον δεν μπορεί να ελέγξει. Τελικά, η νομισματική Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο αν έχουμε έναν επενδυτικό οργανισμό και επενδυτική υπηρεσία που θα επενδύει στις χώρες του Νοτίου του Νότου. Ιδάλω δεν θα μπορέσουμε. Ο κ. Ζεριανόπουλο. Στην Ελλάδα οι διαψεύσει των παραμυθιών ΣΥΡΙΖΑ είναι απανοτέ. Πανηγύριζε για αύξηση ψίχουλα στον κατώτερο μισθό, καταργώντας συλλογικέ συμβάσει εργασία. Οι εκβιασμοί εργαζόμενων να δεχθούν από πλήρη τη μερική απασχόληση και οι απολύσει αυξήθηκαν. Σούπερ μάρκετ καλούν εργαζόμενου να ευλογούν το αφεντικό γιατί παίρνουν 300 ευρώ και όχι μηδέν πανηγύριζε που δεν έκοψε 23η φορά τι συντάξει. σαν μέλο τη οικονομική επιτροπή του κοινοβουλίου ρώτησα τον πρόεδρο του eurogroup κύριο σεντένο μήπω θα περικοπούν και πάλι αν δεν πιαστούν τα πλεονάσματα. απάντηση ολοκάθαρη σιωπή. το ευρωπαϊκό εξάμεινο αποκαλύπτει γιατί. η επιτροπή είναι εδώ και γεμάτη αντιλαϊκά μέτρα. Βασικό στόχο τη Ένωση, η διάλυση τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, επικαλούμενη τη δημογραφική γύρανση αφαιρεί κρατικά κονδύλια από τα ασφαλιστικά ταμεία οδηγώντας τα στις μεγάλες επιχειρήσεις. ανταγωνιστικότητα δηλαδή με συντάξεις ελεημοσύνη δουλειά έως θανάτου με ενεργό γύρανση. για όποιον έχει ιδιωτική ασφάλιση τα αποθεματικά της τζάμπα στις επιχειρήσεις μέσω χρηματιστηρίων. η ευρωπαϊκή ένωση με νεοφιλελεύθερους ακροδεξιούς είτε ψευτοπροοδευτικά μέτωπα όπω του σύριζα μόνο χειροτερεύει και γίνεται πιο επικίνδυνη για του λαού. Κύριε Μπέκερ, 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την συνάδελφο Μάριαν Χάρκιν από την ε, Επιτροπή ε, Κοινωνικών Υποθέσεων ε, για την σημαντική της έκθεση. Να ευχαριστήσω όμως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι ε, κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολύ σημαντική δουλειά που είναι απαραίτητη για τη μεταρρύθμιση των κρατών μελών. Είναι όμως γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ε, και δεν καταβάλουν αρκετές ή, καθόλου προσπάθειες ε, για μεταρρύθμιση. Συχνά αντιμετωπίζουν πήγουσες προκλήσεις όμως και ιδιαίτερα όσον αφορά την βιωσιμότητα των κοινωνικών συστημάτων. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον θα πρέπει να έχει ένα πιο αποτελεσματικό όργανο ε, για υπόμνηση και επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου με δώρα προς τους ψηφοφόρους ε, και ε, με έλλειψη σωστών μεταρρυθμίσεων διακυβεύεται η σταθερότητα των κρατών μελών. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε μικρά αδύναμα κράτη-μέλη, αλλά και σε μεγάλα κράτη-μέλη του Νότου της Ευρώπης. Κύριε Ζουκ, ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φυσικά πρέπει να συμφωνήσουμε με πολλά από τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής. Θα πρέπει να στοχεύσουμε στις επενδύσεις, Φερρυπίν. Αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την περιφερειακή ιδιομορφία. Αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις. Εδώ τονίζουμε, ας πούμε, το ρόλο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πριν από έξι μήνες μιλούσαμε για συστημικούς ε, κινδύνους και ελλείμματα αυτού του μηχανισμού. Γιατί αυτός ο μηχανισμός ε, εφαρμόζεται πολύ επιλεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και άλλες επιφυλάξεις που με ανησυχούν και θα τις τονίσω όσον ούπο. Σας ευχαριστώ κυρία Τόμς. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά έχουμε σημειώσει ως Ένωση βήματα πρόοδου, αλλά η κατάσταση διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την οικονομία σε καλή κατάσταση. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο με σοφές επενδύσεις και μια σωστή φορολογική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη να φροντίσουν για κοινωνική μεταρρύθμιση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στη δημογραφική αλλαγή και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς την οικογένεια πολιτική στέγαση δεν ανήκει στι αρμοδιότητε των κρατών μελών. Ε, σε πολλά κράτη-μέλη όμω είναι πολύ άσχημη η κατάσταση για τι ευρωπαϊκέ ε, οικογένειε. Ε, κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν καθόλου λάβει μέτρα στον τομέα αυτών παρότι από την μελλοντική γενιά θα εξαρτηθεί το μέλλον μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ροζάτη. Ένα λεπτό. συμφωνώ με τις απόψεις ε, διαφόρων συναδέλφων που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι η Ένωση αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Έχουμε οικονομική επιβράδυνση. Για τον... Ε, μπροστά μας έχουμε απρόβλεπτα πράγματα λόγω του Brexit, έχουμε εμπορικού πολέμους και τις επιπτώσεις τους και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα έχουμε θέσει στην Κομισιόν. Οι βασικές ευθύνε ε, όμως τις έχουν τα κράτη-μέλη. Η μεταρρύθμιση των, ε, της αγοράς εργασίας ενθαρρύνει το, τους ανθρώπους να εργάζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Ε, αυξάνουμε το δυναμικό της εκπαίδευσης, την έρευνα και την ανάπτυξη. Και έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε και την κατάσταση των προπολογισμών, δικά σε κάθε, κάθε κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι ευθύνε των κρατών μελών. Ενθαρρύνω λοιπόν την Κομισιόν και τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης ιδιαίτερα να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα στις ειδικέ εκθέσεις αναχώρα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι απέναντι σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτοί ήταν ε, οι ομιλητές που είχαν ζητήσει το λόγο. Φτάνουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Είναι περασμένη η ώρα, γι' αυτό μόνο σε ένα πρόσωπο αναπολιτική ομάδα θα δώσω το λόγο. Κυρία Μάλετσις από Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικές οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Α προσπαθήσουμε στο νέο προπολογισμό να ενθαρρύνουμε τις μεταρρυθμίσει αυτές και να τριπλασιάσουμε τα κονδύλια για τις στρατηγικές επενδύσεις, να ενισχύσουμε την νέα αγορά, να καταρρύψουμε τα εμπόδια, να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Εγώ είμαι αντίθετο στην πρόταση της Κομισιόν. Κατά την άποψη της, το βασικό κριτήριο για αυτά τα μία θα είναι ο αριθμός των κατοίκων. Με αυτόν τον τρόπο δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το βασικό στόχο, ότι πρέπει να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, αναπτυξιακή καθυστέρηση και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και μεγάλες δημοσιο... δημογραφικές προκλήσεις. Και πλήττονται μάλιστα και από τη μετανάστευση. Θα πρέπει να τις βοηθήσουμε αυτές τις χώρες αντί να τις ε, κατακεραυνώσουμε και να ε, προωθούμε έτσι τα προγράμματά μας. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να προωθήσουμε τι επενδύσει ε, και υπεύθυνε δημοσιονομικέ πολιτικέ και μεταρρυθμίσει σοβαρέ είναι οι προτεραιότητε τη Κομισιόν, που πριν από λίγε εβδομάδε δημοσίευσε την αξιολόγηση την, ε, με βάση την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη στα κράτη-μέλη στα πλαίσια του χειμερινού πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, για την Ιταλία το πλαίσιο που σκιαγραφείται είναι αρκετά ζωφερό και επικρίνει την κυβέρνηση Κόντε. Θεωρεί ότι έχει γίνει ένα βήμα προ τα πίσω σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Υπάρχουν ανισορροπίε, ε, υπάρχει μεγάλο χρέο ε, και έλλειμμα και δεν πρόκειται να μειωθεί. Ε, ανισότητες ανάμεσα στο βορρά και στο νότο και τεράστια ανεργία από τις πιο μεγάλες, τεράστια ανεργία των νέων και κίνδυνο να υπάρξει επιμόλυνση σε άλλα κράτη-μέλη. Η οικονομική κατάσταση της Ιταλίας έχει επιδεινωθεί σαφώς. Είναι σαφές ότι η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες χρειάζονται μια αλλαγή ρότας και θα πρέπει να βελτιώσουν τους ε, δημόσιους λογαριασμούς αλλά θα πρέπει να κάνουν μεταρρυθμίσεις γι' αυτός. Η Κομισιόν θα πρέπει να επιμείνει περισσότερο σε αυτές τις χώρες οι οποίες ε, δείχνουν ότι δεν είναι στο ύψος των ε, ευθυνών τους. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ένα σύστημα μέσα από το οποίο η ευρωπαϊκή ένωση κυρίως το συμβούλιο και η κομισιόν παρεμβαίνουν στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών διότι η οικονομική πολιτική δεν έχει καμία σχέση με τις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής ένωσης. ανήκει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και μέσα από το σύστημα του ευρωπαϊκού εξαμήνου αυτό που γίνεται είναι οι βρυξέλλες επί της ουσίας να υπαγορεύουν τη δικιά τους οικονομική πολιτική στα κράτη μέλη. με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν την πολιτική λιτότητας και βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής. έχει άραγε καμιά αρμοδιότητα η ευρωπαϊκή ένωση επί των συνταξιοδοτικών συστημάτων? καμία. και όμως με τις κατευθύνσεις που δίνει διαμορφώνει κλίμα και αν υπάρχουν κυβερνήσεις που ενδεχόμενα αντιδρούν τότε μπαίνουν στην black list των αγορών. είναι λοιπόν ένας τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνουν οι βρυξέλλες σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. καλό θα είναι οι βρυξέλλες να ασκήσουν τις δικές τους αποκλειστικές αρμοδιότητες και να αφήσουν τα υπόλοιπα θέματα να τα ασκούν τα κράτη μέλη και για την πολιτική των μισθών και για την πολιτική των συντάξεων. ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για την ανική ανεργία ε, και τους μισθούς που δεν αυξάνονται αρκετά γρήγορα. Όμως, δεν είναι αυτό να είναι συνέπεια του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά ε, εργασίας με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, εφόσον είναι πολλοί εκείνοι που ψάχνουν ε, ε, εργασία, ε, προφανώς τα πράγματα δυσκολεύουν για τους άλλους που ήδη έχουν δουλειά. Μιλήσατε για την αργή οικονομική ανάπτυξη, αλλά λέτε ότι οι κοινωνικοί σας ε, στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί με την αναπτυξιακή πολιτική. Αν ακολουθήσετε τέτοια προσέγγιση, προφανώς και θα ε, επιβραδύνετε την οικονομική ανάπτυξη. Είναι λογικό. Ο καλύτερος τρόπος να αυξήσουμε το βιτικό επίπεδο, να έχουμε μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα για να μπορέσουμε να τα δαπανίσουμε σε όλα αυτά τα ωραία και θεάρεστα ε, έργα, είναι να αναπτύξουμε την οικονομία με σοβαρές πολιτικές. Κανείς δεν μπορεί να γίνει καλός σομαρίτης αν είναι φτωχός. Αυτοί ήταν οι ομιλητέ στη διαδικασία Καρσιά και τώρα ε, δίνω το λόγο στον κύριο Ντομπρόσκη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, ε, Κύριε εκπρόσωπε τη Προεδρίας, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Θα συνεχίσουμε τώρα το διάλογο με τα κράτη-μέλη και θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοινή κατανόηση των προκλήσεων και των πολιτικών για να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε λοιπόν προγράμματα εθνικής μεταρρύθμισης, τα περιμένουμε μέχρι ε, τα μέσα Απριλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν ε, στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Ε, την ε, Άνοιξη στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα έχουμε τις συστάσεις αναχώρα. Ε, προσβλέπω λοιπόν στη συνέχιση του επικοδομητικού διαλόγου μαζί σας μέσα στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Από το Συμβούλιο η κυρία Τσιώτα έχετε το λόγο παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι, ε, κύριοι επίτροποι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τις παρατηρήσεις σας. Αναφερθήκατε σε σημαντικά θέματα και οι παρατηρήσεις σας ε, θα αποτελέσουν σημαντική συνεισφορά στις συζητήσεις στο Συμβούλιο που άπτονται πολλών πτυχών ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως είναι το περιβάλλον, ε, ο ανταγωνισμός και οι κοινωνικές πολιτικές. Οι εκθέσεις κάθε χώρας που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο αποτελούν σημαντικό βήμα και αποτελούν τη βάση για την δουλειά μας που τελικά θα οδηγήσει στην έκδοση των συστάσεων αναχώρα κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Ε, κατά τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των συστάσεων αναχώρα θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι πρέπει να ε, ε, επικοινωνήσουμε, να έχουμε επαφή με όσο γίνεται περισσότερους πολίτες για να ενισχύσουμε το αίσθημα οικειοποίησης. Η σημερινή συζήτηση έδειξε ότι παρότι υπάρχουν ε, διαφωνίες, υπάρχει και ε, κοινό έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε. Και αυτό με κάνει αισιόδοξη όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τον εντοπισμό των κατάλληλων λύσεων. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Φτάνουμε στους εισηγητέ. Πρώτα δίνω το λόγο στον κύριο Φάντεν Κεντελάρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Το εξάμεινο ανοίγει βεβαίως ε, τις θύρες ε, για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσει και επί της οικονομίας και επί άλλων ζητημάτων. Ε, μπορεί να μην συμφωνήσουμε πάντα για τις προοπτικές, αλλά συμφωνούμε ε, με τους στόχους. Υπήρξαν λοιπόν διαφωνίε και δικαίω. Είναι πολλές οι προκλήσεις, ε, κλιματική αλλαγή, φτώχεια, ανάπτυξη, ανισότητες ε, και γύρανση του πληθυσμού. Όποια και αν είναι η πρόκληση που ακολουθούμε περισσότερο, με βάση τις προσωπικέ μας πεπιθήσεις, Μόνο με τι επενδύσει ή μόνο με την δημοσιονομική πειθαρχία δεν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε ένα μείγμα ε, επενδύσεων, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομική πειθαρχία. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο πρέπει να το κατονομάσουμε ως αυτό που είναι. Μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για τις μεγάλες ε, προκλήσεις που μας περιμένουν. Και βασίζομαι και στη δική σας συμβουλή για την ε, πρακτική υλοποίηση όλων αυτών, ούτω ώστε να το δείτε περισσότερο σαν μία σύσταση και όχι τόσο ε, ως μια τιμωρία που επιβάλλει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε την καλύτερη δυνατή ε, πραγματικότητα στην επόμενη γενιά, στον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ισηγητά για την πολύ καλή σύνοψη αυτή. Κυρία Χάρκινος, εισηγήτρια έχετε δύο λεπτά. Ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να ακούσουμε την εισηγήτρια. Έκθεση δημιουργείται, ε, δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα θα πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη. Θέλουμε και ένα follow-up από την Κομισιόν. Η Επίτροπος Τάισεν ε, χρησιμοποίησε κάποιες από τις προτάσεις της εκθεσής μου. Την ευχαριστώ ειδικά για το θέμα της στόχης και τη ρύθμιση των μεταρρυθμίσεων. Ορισμένες συνάδελφοι μίλησαν για τις συντάξεις. Και φυσικά Θέλουμε καθολική πρόσβαση σε επαρκή σύνταξη και συνταξιδοτικά συστήματα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε και άλλε οδού και μία από αυτέ είναι να συμπληρώσουμε τι υποχρεωτικέ συντάξει με επικουρικέ συντάξει. Τρία τελικά σημεία. Μετά από τη συζήτηση σήμερα για την κλιματική αλλαγή, έχουμε μια τεράστια πρόκληση για, λόγω αυτού του θέματος. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθούν κονδύλια για να απανθρακώσουμε τη βιομηχανία τη ε, μεταφορές και την ενέργεια και να την εξυγχρονίσουμε. Για την κοινωνική ένταξη ζητάμε από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για μεγαλύτερη ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίε στην ε, αγορά εργασία. Λυπούμαστε για την αποτυχία να λάβουμε υπόψη τους αστέγους και τη στέγαση στι προτεραιότητε του 2019. Και ζητούμε από την Κομισιόν να χρησιμοποιήσει αυτό το εξάμεινο για να παρακολουθήσει και να στηρίξει την πρόοδο για φτηνά, φτηνή στέγη, ε, ειδικά σε